Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν από την ε, συνεδρίαση της 6ης Απριλίου είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε θεωρούνται ε,